γιατί εμείς θα έχουμε χρηματοδότηση 85% και όχι 75% και χώρες όπως η Πορτογαλία. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χώρο Σέγγεν και να ορίσουμε προτεραιότητες καθώς και να βελτιωθούμε. Αυτό είναι ένα ε, βήμα αποφασιστικής σημασίας. Ευχαριστούμε κύριε Κόρη. Ευχαριστούμε. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος ε, Πέτερ Μιούλα από τους Σοσιαλδημοκράτες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι κυβερνήσεις αρνούνται το γεγονός, ότι είναι γεγονός όμως, ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Στη σημερινή συζήτηση λοιπόν συζητάμε ακριβώς αυτό το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τους οικονομικούς πόρους. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν να ε, συνεχίσουν να σέρνονται στα θέματα των μεταναστών χρειαζόμαστε τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη. Νομίζω πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους, να μετατεθεί σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να συσταθεί το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική πρέπει να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή και η προστασία των συνόρων δεν ισούται με τις επιστροφές, ε, τις επαναπροωθήσεις, ούτε με το να φυλάσσονται οι άνθρωποι σε καταβλισμού. Πρέπει να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύονται και τα σύνορα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πολύ ωραία. Ε, ο κύριος Βίστησεν για ένα λεπτό. Έχουμε τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις και τις, τη μαζική παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει αποδείξει ότι οι υποσχέσεις για αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα αυτά δεν ελέγχθησαν και δεν τηρήθηκαν στο Σέγγεν. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση και γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρόταση που έχει κατατεθεί λυπούμεθα ε, για το ότι η πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει τα πράγματα σε διαφορετική κατεύθυνση από εκεί που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή έχουμε μετατεθεί από το στοιχείο της ασφάλειας ε, ε, η ομάδα η δική μας, ε, το ECR, δεν μπορεί απλά να παρακολουθεί ε, το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταθέτει τα πράγματα σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε. Ελπίζουμε το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσουν την κατάσταση και να μεταφέρουν την πρόταση στην αρχική της μορφή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίστησεν και τώρα η Μαρή Χριστίν Βεργιά από την ΚΟΕ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγητή που έκανε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνουν αποδεκτά αυτά τα ταμεία, να είναι λιγότερο κακά, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε για ένα οικονομικό ε, εργαλείο της Ευρώπης οχυρό την οποία καταγγέλουμε. Αυτή η λογική της ασφάλειας πάντα βρίσκει χρήματα. Πενταπλασιασμός του, του προπολογισμού 9 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 12 δισεκατομμύρια Frontex, δηλαδή 2% περίπου του προπολογισμού της Ένωσης. Και όλα αυτά για να χρηματοδοτήσουμε τα συστήματα πληροφοριών. Ε, το, το φακέλωμα δηλαδή. Ε, όλα αυτά έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Drones, η αξιωματική σύνδεση που θα βοηθήσουν τι τρίτε χώρε, το μεταναστευτικό τομέα, ιδιαίτερα τη παράτυπε μετανάστευση βέβαια. Εκεί και εδώ τώρα ανησυχούμε. Περαιτέρω ενισχύσει πάνω από τα 12 εκατομμύρια, από τα 12 δι. Εξωτερικοποίηση των συνόρων, ακόμα και αν περιμένει βεβαίω περιορισμένη αυτή και χαίρομαι γι' αυτό. Επίση, 60% των χρημάτων θα, θα διατεθούν στα, χρή, στα κράτη-μέλη, οπότε αναρωτιέται κανεί τελικά πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή πολιτική εδώ. Ευχαριστώ την κυρία Βερζιά. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Μπάτεν από την ΕΝΕΦ, e οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε Αβραμόπουλε, σε αυτήν την ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όντως αυτό το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια, αλλά και αυτή την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενό Ταμείου Διαχείριση ε, των Εξωτερικών Συνόρων. Ένα Ταμείο για τη διαχείριση εξωτερικών συνόρων και την οικονομική χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την διαχείριση τη πολιτική θεωρήσεων. Διότι πρέπει να ενισχύσουμε βεβαίω την ασφάλεια, αλλά να προστατεύσουμε ταυτόχρονα το πιο βασικό στοιχείο τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση, αυτό που εκτιμούν περισσότερο Ευρωπαίοι πολίτε, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δηλαδή. Πολλαπλασιάζουμε επί πέντε, εδώ πενταπλασιάζουμε τα χρήματα για το επόμενο οικονομικο νομισματικό πλαίσιο 2021-2027 και αυτό είναι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουν δηλαδή ότι θα υπάρξει αύξηση της πραγματικής, της απτής αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Δεν είναι δίκαιο όμω να δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση τη ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων τη Ένωση, όταν το Συμβούλιο πραγματικά ε, αντιστέκεται και δεν δέχεται καμία πρόοδο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης και της βοήθειας για τους ε, προσφύγες, για τους πρόσφυγες. Και εκεί φαίνεται και ποιο είναι το ηθικό μέγεθος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία ε, Σεσίλ Κέγγι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο χώρος Σέγγεν είναι ε, ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκλήρωσης. Ε, μία σωστή λειτουργία χωρίς εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Και αυτό σημαίνει έλεγχο και των ε, εξωτερικών συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα βήμα προς τα μπρος, προς μια κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στον ευρωπαϊκό χώρο με βάση το κοινοτικό κεκτημένο και τις ε, ε, διεθνείς μας υποχρεώσεις. Πρόκειται για μία από τις βασικές μας ελευθερίες και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της μη απόθυσης και της ε, μη διάκρισης, τηρώντας το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κιέγκε. Και τώρα ε, περνάμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο αναφερόμενος στην εισήγηση θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ ότι το θέμα των hot είναι κρίσιμο και αυτό φυσικά το γνωρίζουμε όλοι. γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η μόρια έχει ξεπεράσει τα όρια της στη λέσβο όπως επίσης και το hot spot στη σάμο. δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. και όλα αυτά συμβαίνουν παρότι βεβαίως έχουν δοθεί πολλά χρήματα από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης γι' αυτό και είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος διότι το πάρτι δυστυχώς συνεχίζεται. από εκεί και πέρα θα ήθελα να θέσω και το θέμα κύριε αβραμόπουλε της φύλαξης των συνόρων στην ε, ήπειρο στα ελληνοαλβανικά σύνορα διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει παρουσία της frontex. παρά τα αυτά συνεχίζονται δυστυχώς οι παράνομες είσοδοι κακοποιών από την πλευρά της αλβανίας έχουν ρημάξει κυριολεκτικά τα χωριά και νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε ένταση της φύλαξης να υπάρξουν θερμικές κάμερες και βεβαίως να υπάρξει και συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές γιατί συμβαίνουν και τελωνειακές απάτες. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο Μαριά και τώρα ο Επίτροπος, ο κύριος Αβραμόπουλος, έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αν και σε προκεχωρημένη ώρα, σχετικά με τα θέματα της υποστήριξης των εξωτερικών συνόρων. Ε, το να διευκολύνουμε τα, τις μετακινήσεις, τα ταξίδια και να έχουμε και ασφάλεια στην περιοχή Σέγκεν, αυτό είναι η βασική ε, ανησυχία των πολιτών μας και ακριβώς αυτό είναι και η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πλέον έχουμε επιδείξει την αποφασιστικότητά μας να δραστηριοποιηθούμε σε αυτή την προτεραιότητα διασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση για αυτή την πολιτική και συστήνοντας ένα ταμείο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Και προσβλέπω βέβαια στο να συνεχίσω τη συνεργασία μαζί σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Και τώρα... Τελειώσαμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο θα ψηφίσουμε επί του θέματος. Τώρα ξεκινάμε το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Πρόκειται για το, ε, το Εσωτερικό Ταμείο Ασφάλειας. Ε, θα μας παρουσιάσει την έκθεση η κυρία Χολμάιερ. Ταμείου Ιστορικής Ασφάλειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Φτάσαμε επιτέλους ε, στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης. Είμαστε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και θα ασχοληθούμε με την ιστορική ασφάλεια και με το νέο ταμείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδη ηγητές, οι οποίοι μείναν οι μόνοι που έμειναν εδώ μαζί μου, μαζί με τον κύριο Επίτροπο, ε, για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αυτό το ε, Ταμείο της Εσωτερικής Ασφάλειας αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της ε, απειλής από τη διεθνή τρομοκρατία, όπως επίσης και λόγω της ε, αντιμετώπισης της ε, τρομοκρατίας και τα κρατημέλη καταλήγουν όλο και περισσότερο στην άποψη ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά, ότι θα πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ότι θα πρέπει να συντονιζόμαστε και επίσης ότι ε, πρέπει ε, να είμαστε τεχνολογικά προετοιμασμένοι για όλες τις απαντήσεις. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει το νέο ε, κανονισμό. Εγώ τον θεωρώ μια πολύ καλή βάση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Ως Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε από κοινού με μεγάλη πλειοψηφία να ασχοληθούμε με τα βασικά θέματα, κυρίως όσον αφορά με την βελτίωση της ανταλλαγής ε, πληροφοριών ε, ανάμεσα στις ε, ποινικέ αρχές, καλύτερη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε τις ε, διοκτικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται για θέματα οργανωμένου εγκλήματος ακόμα και όταν υπάρχει η διασυνοριακή διάσταση του εγκλήματος αυτού. Πρέπει να προλαμβάνουμε τα βαριά εγκλήματα, την τρομοκρατία, τα κύβερνο εγκλήματα. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές ε, αλλά και τους ιδιώτες ε, στα κράτη-μέλη. Έχουμε καθορίσει ορισμένα όρια. Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι χρειάζεται πολύς χρόνος μέχρι τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να ανακαλούν τα κονδύλια και να εξετάζουν ε, και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα. Νομίζω ότι οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμάς ε, λόγω του μεγέθους ε, της πρόκλησης. Περιμένουν λοιπόν από εμάς ότι πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά με τα θέματα. Να μην αποτυγχάνουμε στα εθνικά σύνορα. Να μην είναι αυτός ο λόγος που μερικές πληροφορίες δεν δίδονται περαιτέρω, που δεν φυλάσσονται κάποια δεδομένα ή ε, που, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε στο τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Και γι' αυτό το λόγο ε, τολμήσαμε κάτι που ίσως είναι και ασυνήθιστο. Δηλαδή, λέμε, επιθυμούμε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες, μυστικές ε, υπηρεσίες πληροφόρησης. Γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο λόγω της ε, τρομοκρατίας να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών στις μυστικές ε, υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση η Europol μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να δημιουργεί ένα δίκτυο για να μπορεί να αναλύει πληροφορίες. Αν λοιπόν θέλουμε να διευρύνουμε την Europol είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να είναι προσαρμοσμένα στο να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Όμως θέλουμε να πούμε επίσης με απόλυτη σαφήνεια ότι και ο ιδιωτικό τομέας μπορεί να ενταχθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο και μπορεί να γίνει αποδεκτός βέβαια με κάποιους περιορισμούς. Ο ιδιωτικό τομέας ε, δεν είναι βέβαια ε, αρμόδιος, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση του ιδιωτικού τομέα ε, για τέτοια θέματα που συζητάμε μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Μόνο τότε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ιδιωτικό τομέας όταν έχουμε να κάνουμε με ασφάλεια, με τράπεζες. Εκεί πράγματι ε, πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία. Αλλά το να αναλαμβάνει ο δυτικό τομέα ε, δημόσια καθήκοντα νομίζουμε ότι δεν είναι σωστό. Αυτά τα καθήκοντα θα πρέπει να παραμένουν στα χέρια των εθνικών αρχών ασφαλεία. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία και με τρίτε χώρε Να συνεργαζόμαστε με ε, τους οργανισμούς που είναι σημαντικοί γιατί τη διεθνή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μόνο αν συνεργαζόμαστε και με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έχει το λόγο, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη γρήγορη εργασία προπαρασκευή τη έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια. Σα ευχαριστώ και για την εισαγωγή σα, κυρία Χολμάιρ. Ήδη έχω υπογραμμίσει στις προηγούμενες συζητήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και τα τρία ταμεία. Ανάγκη ευελιξίας, συνέργειας ε, με τα άλλα ταμεία. Όπως είπα, ελπίζω το Συμβούλιο σύντομα να εγκρίνει την διαπραγματευτική της εντολή. Διαπραγματευτική του εντολή. Τώρα θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που αφορούν ε, πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια οι επιλέσεις για την ασφάλεια έχουν αντιδικοποιηθεί και έχουν επίσης ε, ποικίλε μορφές πλέον. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να τα αντιμετωπίσουν μόνα τους. Πρέπει να προστατεύσουν βεβαίω οι πολίτε και αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθοριστικό για τα επόμενα χρόνια και οι, Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν δικαίως από την Ένωση αλλά και από τις κυβερνήσεις τους να μπορέσουν να τους προσφέρουν ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και που διέπεται από ας ανασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικές προτεραιότητες στις οποίες βασίζεται αυτό το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας και βεβαίως έχετε να συμπληρώσει άλλα ταμεία. Προτείνουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τον προπολογισμό για την ασφάλεια από 1 δισεκατομμύριο στην παρούσα περίοδο σε 2,5 δισεκατομμύρια στην επόμενη. Αυτό αποτυπώνει και την πολιτική σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια. Βεβαίω τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται. Γι' αυτό λοιπόν, και πιστεύω ότι εδώ συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό η χρηματοδότησή μα να είναι ευέλικτη να είναι απλή και να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες όταν αυτές αλλάζουν. Πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει καλύτερα το Ταμείο ε, ε και θα σας βοηθήσει για να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις. Θέλουμε να αυξήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, θέλουμε να εντατικοποιήσουμε τις διασυνοριακέ κοινέ επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες καταπολέμησης και πρόληψης του εγκλήματος θα είναι πιο ευέλικτο λόγω της θεματικής διευκόλυνσης και της ενδιάμεσης αξιολόγησης που μας επιτρέπει να διαθέσουμε ε, τα χρήματα με βάση την εξέλιξη των αναγκών. Τέλος, η ασφάλεια είναι ένα οριζόντιο ζήτημα. Αφορά πολλούς τομείς πολιτικής και αγγίζει πολλά ευρωπαϊκά ταμεία. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κάνουμε μια σωστή επιλογή έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει το χρόνο αυτό το ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αβραμόπουλε και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη των ομάδων, η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μόνικα Χολμάιερ, για την ε, κοινή μας εργασία. Τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς απειλές διαφοροποιούνται και οι προκλήσεις ε, δεν μπορούν να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών θα πρέπει να βρούμε μία συντονισμένη απάντηση σε επίπεδο ένωσης καθώς και τους κατάλληλους πόρους για αυτό το τομέα ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Όμως τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο ε, ασφαλείας με πρόληψη, συντονισμό και συνεργασία. Με βάση τους πόρους αυτού του ταμείου, τα κράτη θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και την μυσαλλοδοξία και την ριζοσπαστικοποίηση με μια μεγαλύτερη συνεργασία δημοσίων αρχών και κοινωνίας των πολιτών. Ένα βασικό ζήτημα είναι η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα στα πλαίσια αρχών που ορίζονται από τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση έτσι ώστε να υπάρχει και κατάρτιση του προσωπικού για να μην ε, προωθείτε καμία μορφή ρατσισμού. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κέγγε. Η επόμενη ομιλήτρια από το ECR είναι η κυρία Χέλγκα Στίβενς. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα διευσυνοριακά προβλήματα, ε, η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Γι' αυτό συστάθηκε και αυτό το ταμείο. Για να έχουμε ενσωμάτωση όλων των ε, τραπεζών δεδομένων των κρατών μελών και να χρησιμοποιηθούν και τα εθνικά συστήματα πληροφοριών. Νομίζω ότι θα πρέπει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση αυτού του ταμείου και επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την επιγραμμική παιδεραστία. Επίσης, αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού θα πρέπει να καλύψει και την ασφάλεια των πολιτών. Όμως μερικά κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότηση εάν προσκρούει σε θέματα ιδιωτικότητας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Στίβενς από τους Πρασίνους τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος Ρωμαίο Φραντς για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της σε αυτό το θέμα. Εμείς οι πράσινοι, για λόγους αρχής, είμαστε υπέρ της καλύτερης συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και ε, τώρα έχουμε να ψηφίσουμε για ένα κείμενο που περιλαμβάνει καλούς ε, συμβιβασμούς. Μεταξύ αυτών ε, και το πρόγραμμα Εράσμους έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τις ε, αρχές δίωξης. Εμείς όμως θα καταψηφίσουμε την έκθεση για του εξή λόγου. Πρώτον, προβλέπεται η αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στι ε, μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας και εκεί το Κοινοβούλιο δεν έχει έλεγχο. Το 5% των κρατών μελών ε, ε, ζητούν ε, ε, να δοθούν περισσότερα κονδύλια σε αυτές τις μυστικές υπηρεσίε. Και δεύτερον, θα μπορούσαν να προαχθούν στρατιωτικές πλατφόρμες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Σε τελική ανάλυση για μένα είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στην έκθεση αναφέρεται και η ε, interim crime είναι μία έννοια που πολλές φορές χρησιμοποιείται για να ποινικοποιούνται οι εθνικές, οι εθνοτικές μάλλον μειονότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα από την Ενωμένη Αριστερά η κυρία Κορνέλια Έρνστ. Κυρίες και κύριοι, ε, νομίζω ότι δεν είναι μυστικό το ότι αυτό το ταμείο δεν είναι και το αγαπημένο μας. Ε, Υπάρχουν βέβαια κάποιες βελτιώσεις, το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Αυτό όμως που δεν μας αρέσει είναι πρώτον ε, ότι προβλέπεται μεγάλη αύξηση κατά 1,5%. Το δεύτερο είναι οι περίφημες blending operations, δηλαδή θα περιλαμβάνεται χρηματοδότηση και από ιδιώτες. Επ' αυτού τοποθετήθηκε η συγγήτρια. Για μας όμως αυτό δεν είναι σαφές και γι' αυτό το λόγο ανησυχούμε. Και το τρίτο θέμα είναι και το σημαντικότερο, δηλαδή το ταμείο αυτό θα προάγει τη συνεργασία ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες υπηρεσίε, όπως πολύ ωραία λένε, για να υπάρχει μια κοινή νοοτροπία μυστικών υπηρεσιών, ε, να χρησιμοποιούνται βέλτιστέ ε, πρακτικές. Κοιτάξτε, α το πω ειλικρινά, τουλάχιστον στη Γερμανία, σε εμά ε, δεν υπάρχουν βέλτιστέ πρακτικές που να αφορούν τι μυστικέ υπηρεσίε. Οι μυστικέ υπηρεσίε τα συγκαλύπτουν. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι περισσότερο ένα τμήμα του προβλήματο και όχι η λύση του προβλήματο. Και γι' αυτό θεωρούμε κρίμα τα λεφτά. Ευχαριστώ τον κύριο Έρνστ. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Σόσνιερτς. Ευχαριστώ. Το κείμενο αυτό δεν είναι το, καλύ, το χειρότερο βέβαια σε σχέση με άλλα που υπάρχουν στο Κοινοβούλιο, αλλά έχω και κάποια σχόλια, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Πρώτα απ' όλα η θανατική ποινή. Υπάρχουν μέτρα αυτή τη στιγμή κάπως ξεπερασμένα, όπως το είναι κάποιος κατά της θανατικής ποινής. Όσο θα είστε κατά της θανατικής ποινής, ε, θα υπάρχουν τρομοκράτες. Αυτοί θέλουν να μας σκοτώσουν. Άμα δεν, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε εμείς, θα συνεχίσουμε να τους έχουμε. Προβλέπετε εδώ πολλά χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά τα πετάμε το παράθυρο ουσιαστικά, ε, χωρίς θανατική ποινή. Άρθρο 12 τώρα συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες είτε μιλάμε για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είτε όχι. Ακούστε, εδώ χάνεται η αρχή της αλληλεγγύης. Παραβιάζουμε την αρχή της αλληλεγγύης. Και τέλος το άρθρο 21. Εδώ μιλάμε για δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι φαίνεται θέλουμε ε, να κάνουμε κάποια πράγματα και καλυμμένα. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε τελικά τι κάνετε. Θα πρέπει κάπου να μπαίνει και το λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά που υπάρχει χρηματοδότηση της Ένωσης. Διότι εδώ δεν είναι και το δεν υπάρχει μεγάλη συνέπεια στις δράσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σοσνιέρς. Και τώρα διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαριά, παρακαλώ. Πρόεδρε, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να επικεντρωθεί στο χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως στο διασυνοριακό έγκλημα. είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. εγώ θα ήθελα να προτείνω να υπάρχει μια συνεργασία επιπλέον της ελλάδας με τη βουλγαρία διότι έχει αναπτυχθεί κύριε αβραμόπουλε πάρα πολύ το διασυνοριακό έγκλημα. πέραν του ότι έχουμε πάρα πολλούς παράνομους μετανάστες που έρχονται από τουρκία βουλγαρία και εν συνεχεία στην ελλάδα έχουμε πλέον και σπήρες εγκληματιών και κακοποιών οι οποίοι κυριολεκτικά λιμένονται το κέντρο της θεσσαλονίκης με ληστείες ε, κλοπές και εν συνεχεία επιστρέφουν στη βουλγαρία. πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί. είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. από την άλλη πλευρά όπως υπόθηκε το ταμείο εσωτερικής ασφαλείας δεν θα πρέπει να αποτελέσει και χρηματοδότη της συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών όπως επίσης να μην έχουμε και μια είδους ιδιωτικοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας. αυτά είναι σημεία που πρέπει να τα προσέξουμε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαριά. Και τώρα ε, το λέω δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Τον κύριο Αβραμόπουλο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε για αυτήν την ενδιαφέρουσα και σύντομη συζήτηση ε, για το Ταμείο εσωτερική ασφάλεια. Σημείωσα όλα τα σχόλιά σα και τα τελευταία, και το τελευταίο του κύριου Μαριά και ανυπομονώ να λάβω και την εντολή του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίε μα. Ε, ευχαριστώ πολύ και καλή σε όλους. Όχι εδώ όμως, μην κοιμηθείτε εδώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι εγώ είμαι αρκετά κουρασμένη βέβαια. Ε, πρέπει όμως να ακούσουμε και την εισηγητρία, την κυρία Χολμάιερ. Παρακαλώ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα οι γυναίκες έχουν τον τελευταίο λόγο. Ε, δηλαδή εγώ ε, θα είμαι εκείνη που θα μιλήσω λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Να πω λοιπόν στους συναδέλφους τα εξή. Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ τους και ηγητές, γιατί πραγματικά ε, κατέθεσαν πολλές και επικοδομητικές απόψεις και νομίζω και στις συζητήσεις μας είχαμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Προσπαθήσαμε λιγάκι να τα βρούμε και από κοινού να καταθέσουμε ένα κοινό σχέδιο σχέδιο. Όσον αφορά τις ε, μυστικές υπηρεσίες, ε, θα ήταν λάθος ε, να πιστεύετε ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις μυστικές υπηρεσίες. Μα αυτό δεν μας το επιτρέπει καν η συνθήκη. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, παραδείγματο χάρη με την Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο της τρομοκρατίας βλέπουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες πρέπει να αναλύονται, να εξακριβώνονται και μετά να αποφασίζουμε κατά πόσον θα χρησιμοποιούνται για έρευνες που γίνεται από τις ε, αστυνομικές αρχές. Το θέμα αυτό, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, το είδαμε στην περίπτωση Ριτσίν, όπω είναι γνωστή. Αν δεν είχαμε εκεί τι μυστικέ υπηρεσίε, δεν θα μπορούσαμε να αποκαλύψουμε του δράστε. Άρα, δηλαδή, με τι ε, μυστικέ υπηρεσίε, όπω σα είπα, αυτέ δεν θέλουμε να τι ελέγχουμε, ούτε και να τι προωθήσουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε και να το θέλαμε. Εμεί θέλουμε απλά τη συνεργασία ανάμεσα στι μυστικέ υπηρεσίε. Δεύτερον, στρατιωτικέ επεμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό ε, είναι καθαρά ε, προδιαγεγραμμένο. Δηλαδή, αν στη Γαλλία ή στο Βέλγιο υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία βοήθησαν στην περίπτωση της τρομακρατικής επίθεση. αν μπορούν οι στρατιωτικές δυνάμεις να βοηθήσουν σε τέτοιου είδου περιπτώσεις, τότε ναι. Αλλά ε, όχι με οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ασφάλεια. Δεν μπορούν οι αρμοδιότητες των στρατιωτικών δυνάμεων να επεκτατούν. Ε, ακόμα και ε, σε περιπτώσεις εξαίρεσης νομίζω και εκεί δεν μπορούμε να πράξουμε πολλά. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Αν κάποιος λέει ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το θέμα της θανατικής ποινής, εκεί πραγματικά μου γυρίσει στο μάχη κατά λέξη γιατί υπάρχει ε, η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ε, εγκληματίες με τα ίδια μέσα. Εμείς θέλουμε το κράτος δικαίου, την απάντηση να τα δίνουμε με τους δικούς μας τους νόμους, άρα δηλαδή τα δικαστήρια είναι αρμόδια για να αποφασίζουν για τις ποινές και μετά να ε, αντιμετωπίσουν ανθρώπους αυτούς πάντα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση αύριο. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ξεκινούμε ξανά τη συνεδρίαση αύριο, αύριο Τετάρτη, 13 Μαρτίου, στις 9 το πρωί έως τις 2 και μετά από τις 3 έως την ολοκλήρωση. Και μπορείτε να βρείτε έως το 10 το βράδυ δηλαδή. Ε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στη διάταξη. Καλό βράδυ σε όλους και καλή νύχτα.